Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Εντάξει κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε ξανά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Χωσέ Μπλάνκο Λόπες, ο οποίος ε, είναι ο Υπουργός Μεταφορών της Προεδρεύουσας ε, Ισπανίας και μετά επίσης θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με αυτούς που έχουν τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα δώσουμε λοιπόν ε, τον λόγο στον Προεδρεύοντα για να μας πει τι θα θέλαμε να κάνουμε και μετά θα μας πει η Τράπεζα ότι δεν μπορείτε να κάνει τίποτα γιατί δεν έχετε λεφτά. Εν πάση περιπτώσει όμως, ε, δεν έχει άπειρο χρόνο ο κύριος Υπουργός, πρέπει να γυρίσει στην Ισπανία γιατί τον περιμένει μια ψηφοφορία και επομένως θα του δώσουμε αμέσως το λόγο. Λοιπόν, είναι και μετά το γεύμα, μην μας παρεξηγείτε. Έχετε πάντως το λόγο. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στις 27 Ιανουαρίου όταν είχα ξαναέρθει σας είχα παρουσιάσει τις γενικές γραμμές των δράσεων της Ισπανικής Προεδρίας για την πολιτική μεταφορών. Σας έφερα και ένα έγγραφο με προτεραιότητες, ε, το οποίο αφορούσε στο πρόγραμμα εργασίας ε, του τρίου των προεδιών που μοιραζόμαστε με το Βέλγιο και την Ουγγαρία. Και όπως σας είχα υποσχεθεί, εμφανίζομαι εδώ σήμερα για να σας ενημερώσω για την πρόοδο που έχουμε επιτελέσει μέχρι σήμερα. Στις 12 Φεβρουαρίου έγινε στη Λακορούνια η άτυπη σύνοδος υπουργών στην οποία συμμετείχαν και ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Μικελάνχελ Μαρτίνες, ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κύριος Κάλλας, ε, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του μετά από τον διορισμό του στις 12 ε, ε, Φεβρουαρίου και εκεί συζητήθηκαν τα θέματα βελτίωσης της βιωσιμότητας ε, για την αστική και μητροπολιτική κινητικότητα ακολουθώντας ε, την άγουσα που είχε καθορίσει το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως αποτέλεσμα θα υποβάλουμε ένα έγγραφο συμπερασμάτων υπόψη του ε, επομένου Συμβουλίου Υπουργών τον Ιούνιο στον οποίο θα καθορίζονται οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές ώστε σεβόμενοι την αρχή της επικουρικότητας να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Επιπλέον, στην άτυπη σύνοδο συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας ε, στην αεροπλοεία οι Υπουργοί επανεπιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους για να γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας στον ε, αεροπορικό τομέα και θεωρούμε ότι για να ενισχυθεί η ασφάλεια στον αεροπορικό τομέα στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική η οποία θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θεωρούμε ότι για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πιο προηγμένες τεχνολογικές μέθοδοι και αυτές θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ακριβώς λάβαμε υπόψη την εγκατάσταση στον, στα αεροδρόμια ε, σκάνερ ε, σαν μία από τις ε, δυνητικές λύσεις, σεβόμενη πάντα την ιδιωτική ζωή, την υγεία των προσώπων και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται καταλήλως σε κοινοτικό επίπεδο και να μην υπάρχουν προβλήματα για τους πολίτες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε θετικά διακείμενοι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει ε, στο εγγύς μέλλον μία έκθεση που θα σχετίζεται με τη χρήση αυτών ε, των τεχνολογιών και θα αποτελέσει τη βάση για μία πρόταση νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καθοριστούν κοινοί κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, επισημαίνουμε και την ανάγκη να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας στον αεροπορικό τομέα, τόσο σε διμερές επίπεδο, κυρίως με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά και σε πολυμερές επίπεδο, στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Διότι κυρίες και κύριοι όταν είναι παγκόσμια η απειλή θα πρέπει να υπάρχει και παγκόσμια απάντηση. Όπως γνωρίζετε, στις 17, 15 με 17 Φεβρουαρίου έγινε στη Μαδρίτη ο δεύτερος γύρος δραπραγματεύσεως της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για αεροπορικές υπηρεσίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως συνέχεια της ε, συνεδρίασης που είχε γίνει τον Ιανουάριο στη Ουάσιγκτον και εκεί είχαμε κάποιες σημαντικές προόδους ε, στις διαπραγματεύσεις, ε, κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος, αρμοδιοτήτων και κοινωνικών διατάξεων. Αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ουσιαστικά και σε θέματα τα οποία αποτελούν κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα επενδύσεων σε αεροπορικές εταιρείες και την ε, πραγματική ε, το πραγματικό άνοιγμα των αγορών. Γι' αυτό ακριβώ και συμφωνήσαμε με τον Αμερικανό ομόλογο, με τον κύριο Λαχόπ, για έναν επόμενο γύρο, ο οποίο γίνεται στι Βρυξέλλε σήμερα, για να μα επιτρέψει να προχωρήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Στις 25 ε, και 26 Φεβρουαρίου έγινε στη Μαδρίτη η διάσκεψη για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό η οποία κατέληξε με την έγκριση της δήλωσης της Μαδρίτης και με έναν οδικό χάρτη ο οποίος ε, περιλαμβάνει πάνω από 60 πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το ε, στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πρόγραμμα δράσεων σημαίνει ότι θα γίνει και μια πολύ σημαντική πρόοδος και θα ε, υλοποιηθεί το δεύτερο νομοθετικό πακέτο για τον ενιαίο ουρανό, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα για το 2009-2014. Με αυτό θεωρούμε ότι έχουμε πλησιάσει, προσεγγίσει τον τελικό μας ε, στόχο, έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, το οποίο μας επιτρέπει να ε, ε μειώσουμε τις κλιματικές ε, συνθήκες της αεροπορίας, να έχουμε έναν ενιαίο ουρανό και να βελτιώσουμε και την ασφάλεια στον αέριο χώρο. Και για όλο αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και αυτό το είπα και στους συναδέλφους ε, στο Συμβούλιο Υπουργών που έγινε στις 11 Μαρτίου. Στο Συμβούλιο αυτό ενεκρίθη μια ε, γενική γραμμή προσανατολισμού για ένα σχέδιο κανονισμού για την έρευνα και την πρόληψη ατυχημάτων και δυστυχημάτων στην πολιτική αεροπορία, το οποίο ε, θα περιλαμβάνει τις ε, δεξιότητες των ερευνητών, δίνει μεγάλη σημασία στις ε, συστάσεις ασφαλείας, διευκρινίζει το ρόλο της υπηρεσίας αεροπορικής ασφάλειας και ενισχύει το θέμα της συνδρομής στα θύματα. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το τελευταίο σημείο, διότι όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες να διαθέτουν πληροφορίες ε, για τα άτομα τα οποία βρίσκονται εντός ενός αεροπορικού σκάφους όταν γίνεται κάποιο αεροπορικό δυστύχημα. Δεν θέλουμε να έχουμε ε, μεγάλες περιόδους άγχους και ανησυχίας ε, στον πληθυσμό, καθώς επίσης και αυτή τη μόνιμη πίεση προς τις αεροπορικές εταιρείες για να λάβουμε τις πληροφορίες που αφορούν τις οικογένειες και τους φίλους τους. Γι' αυτό ακριβώς οι Υπουργοί υιοθέτησαν ένα συμβιβασμό μέσω αυτού του κανονισμού να καθοριστεί μία μέγιστη προθεσμία δύο ωρών για να δοθεί στη δημοσιότητα ο κατάλογος των επιβατών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε τρεις επιφυλάξεις τεχνικού χαρακτήρα σε αυτή την πρόταση κανονισμού, αλλά θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Κοινοβούλιο ή δυνατόν κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Κυρίες και κύριοι, επίσης θα ήθελα να σας πω ότι στο Συμβούλιο έγινε και μία ενημέρωση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για την οδηγία για ε, τους... Ε, ε, τα επίπεδα ασφαλεία στην αεροπλοεία. Εκεί έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες για πολύ συγκεκριμένε πτυχές ε, ουσία τη πρόταση. Γι' αυτό ακριβώς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί το εν λόγω κείμενο στο Κοινοβούλιο τον Απρίλιο προκειμένου να ε, συνεχίσουμε τη μελέτη του. Στο Συμβούλιο Μεταφορών επίσης καθορίσαμε κάποιους γενικούς προσανατολισμούς ε, για το σχέδιο οδηγίας για εξοπλισμούς υποπίεση μεταφερόμενους που θα βελτιώσει την ασφάλειά τους και θα διασφαλίσουμε ταυτόχρονα ότι θα υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρξει συμφωνία για τι ε, πράξει εξουσιοδότηση. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Κοινοβούλιο ή δυνατόν και αυτό στη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία. Επιπλέον, να σας ενημερώσω ότι προχωρήσαμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία για, την, ε, ε, για τα ευρω... διευρωπαϊκά δίκτυα. Υπάρχει και η πρόταση οδηγίας για το συστήματα ευφυών μεταφορών και καταλήξαμε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο για τις πράξεις εξουσιοδότησης και τις εκτελεκτιστικές πράξεις και ελπίζουμε όταν το Συμβούλιο κάνει την πρώτη του ανάγνωση, το Κοινοβούλιο να το εγκρίνει σε δεύτερη ανάγνωση και να θεωρήσει ότι είναι οριστικό το θέμα αυτό. Επιπλέον στο Συμβούλιο υιοθετήθηκαν και κάποιες ε, θέσεις σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση κανονισμού που σχετίζεται με τα δικαιώματα των επιβατών ε, των σιδηροδρόμων και των θαλάσσιων ε, μεταφορών και η Ισπανική Προεδρία ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση με το Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει να εγκρίνει την ομοθεσία η οποία θα αυξήσει τα δικαιώματα των χρηστών αυτών των μέσων μεταφοράς επισημένοντας κυρίως ε, όλου, ε, ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, σε άτομα με αναπηρία και με μειωμένες δυνατότητες μετακίνησης. Τέλος να σας πω ότι το Συμβούλιο Μεταφορών ενέκρινε και την κοινή θέση για τις προτάσεις ε, απόφασης και σύστασης που υιοθετήθηκαν το 2003 από την Κοινή Επιτροπή Interbus, που σημαίνει ότι έχει γίνει ένα βήμα περαιτέρω για την ε, ε, συμφωνία αυτή που είναι υπέρ της απελευθέρωσης των μεταφορών με τρίτες χώρες και την επέκταση των και, κοινωνικών και τεχνικών κανόνων για τα θέματα αυτά. Κυρίε και κύριοι, όπως θα διαπιστώσατε, το θέμα της αεροπορίας ήταν κυρίως αυτό το οποίο ε, μας απασχόλησε κατά το πρώτο τμήμα του εξαμήνου. Ε, προχωρήσαμε στα θέματα των δυστυχημάτων του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, προωθήσαμε τη βιωσιμότητα με τη συζήτηση που έγινε στη Λακορούνια και προχωρήσαμε και τα νομοθετικά προγράμματα τα οποία θα βελτιώσουν τα ε, δικαιώματα των επιβατών σε λεωφορεία, σε σιδηροδρόμους και σε ε, σκάφη. Αυτά όλα συνάδουν με το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας σε θέματα μεταφορών και θα ήθελα μεταξύ των όσων κάνουμε να σταθώ ε, στο ε, πρόγραμμα το οποίο αφορά στις γενικές μεταφορές το οποίο έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να προχωρήσει η συζήτηση για τα κριτήρια, τη μεθοδολογία της αναθεώρησης οργανώνουμε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία διάσκεψη η οποία θα γίνει στις 8 και 9 Ιουνίου στη Σαραγώσα. Και εκεί θα συμμετέχουν υπουργοί τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από γείτονε χώρε, καθώ επίση και υπεύθυνοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέλη του Κοινοβουλίου. Η συνάντηση αυτή θα μα επιτρέψει να αναλύσουμε το παρόν και το μέλλον των ε, διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Ε, με ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τη μεθοδολογία του καθορισμού του βασικού δικτύου, του RTT, ε, την στρατηγική μέθοδο χρηματοδότησης και τους μηχανισμούς προσανατολισμού και συντονισμού των ε, προγραμμάτων που θα αποτελέσουν προτεραιότητα. Και επίσης εξετάζουμε το ρόλο των διευρωπαϊκών ε, δικτύων ως μέσο που θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε και χώρες γείτονες Ευρωπαϊκής Ένωσης το αποτέλεσμα του Συμβουλίου Μεταφορών του Ιουνίου, καθώς επίσης και τα όσα θα επιτύχουμε στα υπόλοιπα θέματα στους επόμενους μήνες, ε, θα αποτελέσουν αντικείμενο ενημέρωσης όταν θα έρθω τον Ιούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Minister, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ και να θυμίσω ότι παρατέταρτο πρέπει να φύγει ο υπουργό, το λέω για αυτούς που έφτασαν αρκοπορημένοι. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μην κάνετε μεγάλες πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά απλά να θέσετε ερωτήματα. Ο κύριος Γκρός πρώτα και θα έχω πάντα το σφυρί μου έτοιμο να χτυπήσω όταν περάσει ο χρόνος σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ε, βρίσκω πολύ καλό που υποσχεθήκατε να έρθετε και ήρθατε πραγματικά πάλι εδώ. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω στο θέμα των ε, μεταφορών. Ξέρετε ότι πήγε μια μικρή αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον, αλλά παρέμεινα δύο ερωτήματα σημαντικά για μας ανοιχτά. Πρώτον, είπατε ότι υπάρχουν πρόοδοι στον ανταγωνισμό δεν βλέπετε εσείς μια συμφωνία. ώστε να παραμείνουμε σε αυτή την 24% ε, συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ή λέτε ότι θα γίνει κάτι το διαφορετικό. Δεύτερον, ανταλλαγή πληροφοριών. Το SWIFT, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Προσεχώς θα έχουμε μια νέα σημαντική εμπειρία στον ίδιο τομέα. Πώς βλέπετε στη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ούτω ώστε να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, για να το πω έτσι, όπως αυτή του παρελθόντος. Τρίτη, για το σκάνινγκ, για τους ε, σαρωτές σώματος. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον για μας αυτό, πολύ σημαντικό. Παρακολουθήσαμε πώς εξελίσσεται η τεχνολογία και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο το Συμβούλιο θεωρεί ελεύθερη τη χρήση για όλα τα αεροδρόμια ή πώς διαβλέπει την τεχνολογική εφαρμογή και τι γίνεται όσον αφορά την προστασία της υγείας. Όσον αφορά τα τέλη για την ε, ασφάλεια των ε, πτήσεων, χαίρομαι που υπάρχει πρόοδος όπως είπατε, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν διευκρινίσετε την πιο σημαντική ερώτηση. Ποιος προτίθεται να πληρώσει τι δηλαδή και όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, ταξιδιωτών, αυτό κατά τη γνώμη μας είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι στη δεύτερο ήμιση της ε, ε, θήτειας σας θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στο θέμα των οδικών και ιστορικών μεταφορών. Μία ερώτηση μόνο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Η συνάντηση αυτή στη Σαραγκώσα, στην οποία αναφερθήκατε, θα ήθελα να ξέρω εσεί ως Προεδρία Πώς δεν βλέπετε τα πράγματα, δεν βλέπετε νέα κριτήρια, νέες ιδέες να αφορά τη χρηματοδότηση. Ή και διαφορετική συγκριτική αξία των διαφόρων σχεδίων. Και θα ήθελα εδώ να παρατηρήσω, γιατί τα πρώτα δύο σημεία ήταν τα πιο σημαντικά, να μην έχουμε πάλι ένα νέο κατάλογο νέων προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ. Από τους ε, σοσιαλιστές, ο κύριος Αλκαδράουι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τα όσα μας είπατε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και βεβαίως χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε συχνά κοντά μας και εκτιμούμε τη δέσμευσή σας αυτή όσον αφορά τώρα τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω ότι θα στεφθεί από ε, επιτυχία όπως ε, τουλάχιστον είπαν και οι συνάδελφοι που πήγαν την προηγούμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γεγονός ότι ούτως γεγονό θα πρέπει ούτω η πρώτη φάση διαπραγμάτευσης και θα ήθελα την άποψή σας. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η φάση σύντομα. Επίσης, ε, όσον αφορά δύο σημεία τα οποία για μας είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα είναι και τα πιο δύσκολα, η πρόσβαση στην αγορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ αφενός και αφετέρου ε, η διαφάνεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, διαφάνεια όσον αφορά ας πούμε, την απαγόρευση των ε, νυχτερινών πτήσεων στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι πρώτες ερωτήσεις μου. Αλλά και κάτι άλλο υπάρχει που είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως δεν είναι το τέλος για μας. Υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία άπτονται των αεροπορικών μεταφορών επί των οποίων θα πρέπει και να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Είναι πάρα πολλά τα σημεία αυτά ε, που οπωσδήποτε ε, θα μας απασχολήσουν μετά από την ε, συμφωνία αυτή. Safety and security. Πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά τα οποία σχετίζονται με ενεργητική παθητική ασφάλεια. και επίσης ε, τα κέντρα συντήρησης είναι πολύ σημαντικά. Γιατί ακούσαμε και στο Κογκρέσο να συζητούνται πράγματα τα οποία δεν μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνος. Αυτά όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές. Άλλο θέμα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TNT. Περιμένουμε βεβαίως τι θα γίνει και στη Σαραγώσα. Ε, συναντώνται διάφορες ομάδες εργασίας, συζητούν το θέμα αυτό. Κατανοούμε βεβαίως ότι η συνέχεια της συζήτησης δηλαδή η μελλοντική συζήτηση θα πρέπει να συνδεθεί με, την, ε, με το γενικότερο μέλλον των μεταφορών. Μπορείτε να μας πείτε κάτι και να μας πείτε και τι ε, σκέφτεται και το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κυρία Ελκαντράου Η κυρία Ντιλμπά από τους φιλελεύθερους. Τρία λεπτά παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και ευχαριστώ τον Υπουργό για όλες τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Εγώ θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσω κάποια πράγματα και να εστιάσω σε μια αναφορά που κάνατε για την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών μεταφορών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα, διότι διαβάζουμε και ακούμε ειδήσει για την γραμμή προτεραιότητας 3, για μια νέα συμφωνία της γαλλικής κυβέρνησης, μέσω της οποίας τροποποιείται το πρόγραμμα αυτό για την γραμμή προτεραιότητας ε, στο γαλλικό κομμάτι. Θα ήθελα να ε, μάθω κατά πόσον αυτή η νέα διαδρομή που διαβάζουμε στις ε, Ε, στις, ε, στον τύπο θα περάσει και από το Σαν Χουάν Τελούθ και θα δώσει μια νέα γραμμή ταχείας ε, μεταφοράς. Ισχύει αυτή η είδηση που μάθαμε, είναι σωστές οι πληροφορίες και αν όντω είναι σωστές οι πληροφορίες μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Αν υπάρχει ήδη συμφωνία με την γαλλική κυβέρνηση για την εκτέλεση αυτής της γραμμής προτεραιότητας, αν υπάρχει συμφωνία, τι προθεσμίες έχετε προβλέψει και γιατί τροποποιήθηκε αυτό το κομμάτι της διαδρομής. Όσον αφορά στη διάσκεψη που μας αναφέρεται για τις 8 και 9 Ιουνίου στη Σαραγώσα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για τη μεθοδολογία που θα καθορίσετε σε αυτή τη διάσκεψη για τα βασικά δίκτυα, το νέο σύστημα χρηματοδότησης, καθώς επίσης και το συντονισμό των προγραμμάτων προτεραιότητας. Τα αναλύετε, έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση την οποία θα παρουσιάσετε για αυτές τις τρεις πτυχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που δεν ξεπεράσατε το χρόνο σα, Ο κύριο Κρέμερ από του πράσινου. Ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε εδώ για να μας παρουσιάσει την έκθεση για την ε, ασφάλεια των αεροπόρων μεταφορών. Θα έχω να υποβάλω μια ερώτηση, αλλά θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Η νέα μορφή των διευρωπαϊκών δικτύων. Καλά ακούγεται, πήραμε και την απόφαση. Η προτεραιότητα είναι για να ε, αρθούν τα με των τονοπές που υπάρχουν, δηλαδή με τα νέα χρήματα να υπάρχουν γλίγορα ε, αποτελεσματικά, ε, σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της προστασίας του κλίματος και στην επιτάχυση των μεταφορών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ορισμένα από τα σχέδια αυτά που θα ετοιμαστούν σε 20-30 χρόνια από τα μεγάλα αυτά σχέδια και όταν δούμε τα σχέδια που υπάρχουν για τη σύραγγα κάτω από τον Μπρένερ ή ε, το, η σύραγγα Λιον Τουρίνο, άμα από αυτά τα, τα καταφέρουμε σε 30 χρόνια δεν θα έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να λήξουμε τώρα ε, την ε, άγουσα για την βινιέτα, για το ΣΥΜ αυτό το ευρωπαϊκό. Δεν αναφέρατε τίποτα. Η Ισπανική Προεδρία στην αρχή είχε πει ότι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνανε οι ε, προκάτοχοι, δηλαδή να το αφήσουν κατά μέρο, αλλά θέλουν κάτι να κάνουν. Υπάρχει στραβή του νομισμού αυτή τη στιγμή ε, στην Ευρώπη λόγω αυτού. Εσείς θα κάνετε κάτι ή θεωρείτε ότι δεν έχετε καμία πιθανότητα επιτυχίας. Τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα των ταξιδιωτών στα λεωφορεία, στα τρένα, στα πλοία κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει βέβαια κα... κατανομή, παραδείγματο οι δρομικές μεταφορές. Έχω μετά από μία ώρα καθυστέρηση 25% ε, επιστροφή, δύο ώρες καθυστέρηση 100% επιστροφή του τιμής του εισιτηρίου. Στις αεροπορικές μεταφορές μετά από τρεις ώρες έχω δικαιώματα ως ταξιδιώτης. Δεν πρέπει να γίνει και εκεί κάτι για να μην υπάρχει στρέβλωση στον γνωστό. Η ηλεκτρονική ή e-mobility, δεν την αναφέρεται καθόλου κύριε Υπουργέ. Όσον αφορά ε, αυτό το τομέα εννοείται μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή και ηλεκτρικά ποδήλατα, λεωφορεία, τρένα και εκεί μπορούμε να προστατεύσουμε το κλίμα σίγουρα. I still have to speak. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα πολλούς, έξι αγορητές στον κατάλογό μου. Και λοιπόν θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ζήλε, Τούσας, Αλβέιρα, Λίχτεμπερ και κυρία Σάντα. Α, κυρία Μάισνερ. Και δεν δέχομαι κανένα άλλο όνομα, γιατί όπως σας είπα πρέπει να φύγει σε λίγο ο κύριος Υπουργό. Ακόμα και να σηκώσετε τα χέρια σας θα τα αγνοήσω τώρα. Ζήλα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό για τα όσα μας είπε όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας. Η ερώτησή μου αφορά θέματα τα οποία έθιξε ο κύριος Γκρός προηγουμένως. Ε, οι εισαρωτές σώματος με απασχολούν. Ε, έχουν γίνει μελέτες όσον αφορά παρόμοια ενδεχομένως μηχανήματα, ε, υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι, εναλλακτικοί τρόποι ελέγχου ασφαλείας. Θα ήθελα να μου μιλήσει για το θέμα αυτό ο κύριος Υπουργός όσον αφορά τη διάσκεψη της Αραγώσας. Είπαμε ότι θα γίνει λόγος και για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος χρηματοδότησης ε, των δικτύων αυτών. Το Συμβούλιο και οι Υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν το θέμα αυτό από όσο ξέρουμε και βλέποντας το πολύ εγγύης ε, μέλος, μέλλον, βλέποντας ε, και την οικονομική κατάσταση σε χώρες μέλη και όσον αφορά και την δυνατότητα χρήσης ε, του Ταμείου Συνοχής για μεγάλα έργα, οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι χώρες οι οποίες έχουν δύσκολα από απόψεως προγράμματα θα έχουν δυσκολία εφαρμογής των των προγραμμάτων και ίσως θα πρέπει να τα ξεχάσουν αυτά τα προγράμματα, τα TNT. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τούσας. Η υλοποίηση και η πρόοδος της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, χερσαίες, εναέρες και θαλάσσιες, κρίνεται το κατά πόσο συμβάλλουν στην ανάπτυξη, συμβάλλουν κατά πόσο βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς και στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Ε, χρειάζεται να επισημάνουμε ότι σε αυτή τη φάση στις αεροπορικές εταιρείες στην British Airways ε, υπάρχουν μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις γιατί έχουν εξαγγελθεί μαζικές απολύσεις και με τις περικοπές. Ε, το προηγούμενο διάστημα ήταν στην ε, πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία στην Ελλάδα και είναι σε φάση κινητοποιήσεων, έχουν εξαγγείλει απεργιακέ κινητοποιήσει στη Λουφχάνσα. Είναι προφανέ ότι οι συνέπειε είναι πολύ επώδυνε ό,τι αφορά στου εργαζόμενου, αλλά και το οικονομικό βάρο ό,τι αφορά στου χρήστε. Δεύτερο στοιχείο. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μα, είναι επαχθής σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικονομικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των επιβατών και την υγεία των χρηστών. Άρα και είναι και ένα δεύτερο σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά τις συνέπειες που έχει συνολικά για τους εργαζόμενους στα κράτη-μέλη. Και το τρίτο στοιχείο που θα ήθελα είναι το εξής. Η παράμετρος η μία έχει το κατά πόσο οργανώνει η αεροπορική εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά την ασφάλεια, τα επίπεδα ασφάλειας της αεροπλοείας. Κύριε Υπουργέ, έχει διαπιστωθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Αιγαίο Πέλαγος πολλές φορές σε, καθημερινά, σε καθημερινή βάση παραβιάζεται ο εναέριος χώρος, ο ελληνικός, από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που αυτό εγκυμονεί κινδύνους τόσο σε ό,τι αφορά την αεροπλοεία. Ήδη πριν λίγες μέρες ε, υπήρξε κίνδυνος να καταρριφθεί ελικόπτερο της Frontex που περιπελούσε στην περιοχή. Πώς αξιολογείται αυτές τις παρεμβάσεις όταν με τεκμηριωμένα στοιχεία η ελληνική κυβέρνηση έχει, αποδείξει ότι παραβιάζεται ο εναερίο χώρο και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό σε ό,τι αφορά γενικότερα του κανόνε ασφάλειας αεροπλοείας. Καταδικάζεται αυτές τι παραβιάσεις. Κυρία Άλβαρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και νομίζω ότι μιλάω και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων που με συνόδευσαν στην αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας. Μπορέσαμε εκ του σύνεγγυς να δούμε πόσα πολλά προσπαθεί να κάνει η Ισπανική Προεδρία για τις μεταφορές, κυρίως σε μια τόσο δύσκολη στιγμή όπως είναι η τωρινή. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο αναφέρεται και εδώ θα εστιάσω και την απάντηση, ερώτησή μου. Αναφέρατε μια συνεδρίαση υψηλού επίπεδου στο Μόντρεαλ. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της Προεδρίας και ποια θα είναι η τοποθέτησή σας ε, για την ε, λειτουργική ασφάλεια σε ένα τομέα ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεν μπορούμε να ρίξουμε τις αμυνές μας. Επίσης θα ήθελα να αναπτύξετε λίγο περαιτέρω αν μπορείτε ε, πώ έχει τρέξει ο κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τι αεροπορικέ υπηρεσίε με τι ΗΠΑ, για τη συμφωνία με τον ανοιχτό ουρανό που όπως είπατε και εσείς ε, σήμερα ξεκινά ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα βασικά ε, προβλήματα, οι βασικές προόδοι και τι πιστεύετε εσείς ε, ως προς το κατά πόσο θα επιτύχουμε συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας για το, για, τον, για το χρονικό αυτό διάστημα και όντως είναι πολύ φιλόδοξο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ βεβαίως η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και από αυτού θα ήθελα να σας ε, κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ε, ε, ερωτήσεις βεβαίως επί των οποίων θα πρέπει κάπως να απαντήσετε. Πρέπει να βρούμε απαντήσεις για τα θέματα αυτά, γιατί διαφορετικά δεν θα λύσουμε τίποτα. Η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση βασίζεται σε πάρα πολύ περιορισμένους πόρους. Επομένως θα πρέπει να ξέρουμε ποιος θα χρηματοδοτήσει τι και πόσο. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σε σχέση με τα αεροδρόμια, τον αριθμό των επιβατών και τα λοιπά. Γιατί διαφορετικά ε, τα πράγματα δεν είναι σαφή. Και βεβαίω εδώ γίνεται λόγο μονάχα για τα εμπορικά αεροδρόμια. Επίση, θέλω να ξέρω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνουν ε, δεκτές σε αυτή τη διαδικασία ομάδες επιβατών ε, που ενδεχομένως θα αυξήσουν το κόστος ασφαλείας των αεροδρομίων. Όπως είπα και προηγουμένως, το πρόγραμμα μου φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξο. Όμως πρέπει να σκεφτούμε όλοι επί ορισμένων ε, ε, θεμάτων και όχι διαρκώς να αφήνουμε για αργότερα κάποια ζητήματα όπως ας πούμε το θέμα των σαρωτών σώματος. Είμαστε βέβαιοι ότι με τα σκάνερ θα έχουμε καλύτερη ασφάλεια και επομένως ε, φτάνω στην ε, συγκεκριμένη ερώτηση. Έχουν γίνει κάποιες προσωμιώσεις ε, έτσι ώστε να ξέρουμε κατά πόσον θα βοηθήσουν πραγματικά τα σκάνερ στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Um, Ευχαριστώ πολύ. Δύο σύντομα ερωτήσεις έχουμε μόνο πάνω σε αυτά που μας είπατε. Πρώτον, όταν πρόκειται να προετοιμάσουμε μία απόφαση για την χρήση των σαρωτών σώματος. Εσείς θα ζητήσετε να είναι υποχρεωτικά σε, ένα, σε κάποιο αεροδρόμιο ή θα ζητήσετε ότι αυτό θα αφορά μόνο εκείνους που το εισάγουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Δεύτερον, όσον αφορά την αναθεώρηση των ΤΕΝ, των διευρωπαϊκών δικτύων είχαμε εδώ μια έντονη συζήτηση που συνεχίζεται. Σας ρωτώ, εν ώψη των οικονομικών προβλημάτων των κρατών μελών, δεν, θα πρέπει να σταματήσει η εργασία στα διευρωπαϊκά δίκτυα βέβαια, αλλά θα πρέπει ορισμένα μεγάλα σχέδια να τα ξανασκεφτούμε, να τα αναβάλουμε ενδεχομένω ε, θεωρείτε ότι αυτό είναι βατό ή θέλετε να βασιστείτε στα μεγάλα παραβλέποντας τις βελτιώσεις στα μικρά. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις πρόοδους που έχετε επιτύχει μέχρι τώρα για τα θέματα των δικαιωμάτων των επιβατών στο θαλάσσιο τομέα. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να επεκταθεί και ε, κυρίως για ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικότητας και να αποτελέσει και το μοντέλο για βελτίωση σε άλλους τομείς που έχουν πιο ε, παροχημένη νομοθεσία. Ε, όσον αφορά στη διάσκεψη της Μαδρίτης, ε, στην οποία μπόρεσα να συμμετάσχω, θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο συστήνετε εσείς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δήλωση της Μαδρίτης. Δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει, διότι τότε όλοι οι φορείς ε, είχαν ενθουσιαστεί με τις δυνατότητες ανταλλαγών που προσφέρονται, αλλά θα ήθελα να ξέρω κάποια επιπλέον στοιχεία. Και τελευταίο, μία παράκληση. Πριν από κάποιες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ε, πολιτική για το 2020, μία πολιτική που θα αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα οικοδομήσουμε, ελπίζω, τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Ο κύριος Κάλλας παρά το γεγονό ότι φοβόμασταν ότι οι μεταφορέ δεν θα είναι και τόσο πολύ ε, παρούσε, μα διαβεβαίωσε ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα ήθελα να ξέρω κάποια πράγματα για τι μεταφορέ για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020. Μήπω ε, τον Ιούνιο η Ισπανική Προεδρία θα μπορούσε να προτείνει στα κράτη-μέλη μία ανταλλαγή απόψεων για το ρόλο των μεταφορών, για να ενισχύσουμε λίγο και την προβολή των μεταφορών στι ε, πιο σημαντικέ προτεραιότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίπεδο. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Υπουργέ. Έχω δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. Η μία αφορά την εναρμόνιση και την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά, ιδίω στι δραματικέ μεταφορέ. Πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν, το ξέρουμε. Και να ρωτιέμαι ποιε είναι οι δυνατότητε που διαβλέπετε για να κινηθεί, παραδείγματο, η Γαλλία προ ένα άνοιγμα Ξέρω δεν είναι εύκολη αυτή η ερώτηση. Θα με διαφέρει το αποτέλεσμα πάντως. Το δεύτερο, αυτή τη στιγμή οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για όλη την Ευρώπη από τη μια άκρη στην άλλη στο διαδίκτυο. Και μια τρίτη ερώτηση, πάλι για τους ερωτές ε, σώματος ε, και γενικά την ασφάλεια στις μεταφορές. Είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να έχουμε ενιαία προσέγγιση. Όλα τα κρατη να προσπαθήσουν να ενδυναμώσουν την ασφάλεια στους ε, αερολιμένες. Το πιστεύετε αυτό επίσης ή νομίζω ότι είναι λογικό η μία να έχουν σαρωτές και άλλοι να μην έχουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία Υπουργέ, υπάρχουν διάφορα θέματα. Από τα body scan ξεκινήσαμε, στα body scan καταλήξαμε. Αν μπορείτε λοιπόν να προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των βουλευτών, θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες. Eh, Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας κάνω μια επενθύμηση. Δεν έρχομαι εδώ για να σας εξηγήσω τους στόχους της Ισπανικής Προεδρίας. Αυτό το έκανα τον Ιανουάριο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσετε ότι πολλά από τα θέματα που θέσετε σήμερα τα έχετε ξαναθέσει τον Ιανουάριο και δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Η απάντηση είναι η ίδια και ο στόχος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς ε, και τα ανέφεραν κάποιοι ευρωβουλευτές. Εγώ ήρθα εδώ για να σας παρουσιάσω ένα ισοζύγιο των όσων έχουμε επιτύχει μέχρι το πρώτο ε, Συμβούλιο Μεταφορών όπως είχα δεσμευθεί ότι θα κάνω όταν ήρθα την πρώτη φορά και τον Ιούλιο θα έρθω για να κάνω μια συνολική επισκόπωση των όσων κάναμε σε θέματα ε, μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Πρώτον, τέθηκε ένα θέμα το οποίο επαναλήφθηκε αρκετές φορές, ε, το θέμα των σαρωτών σώματος. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι έχω την ικανοποίηση να σας πω ότι 27 συμφωνήσαμε στη συνεδρίαση της Λακορούνια ότι το καλύτερο προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια περνά από μια κοινή στρατογική την οποία θα έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συνολική απάντηση για μια ε, παγκόσμια απειλή δεν ε, είναι μένη μεμονωμένη απάντηση για κάθε κράτος μέλος και σε αυτό συμφωνούμε όλες οι χώρες μέλη. Ακόμα και οι χώρες οι οποίες ε, με κάποιο πειραματικό τρόπο έχουν ήδη εντάξει τους αρωτές σώματος, τους αερολιμένες τους. Ω συνέπεια αυτής της συζήτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εκπονήσει μία έκθεση προκειμένου στο Συμβούλιο του Ιουνίου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να λάβουμε μία απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα ετοιμάσει μία έκθεση, θα την παρουσιάσει τον Απρίλιο και εκεί θα αναλύσουμε τις τεχνικές, οικονομικές ε, πτυχές ε, και την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών, την ιδιωτική του ζωή, την υγεία τους και ούτω καθεξής αλλά ταυτόχρονα θα πρόκειται και για ένα κείμενο το οποίο θα χρησιμεύσει για να λάβουμε μια κοινή απόφαση επί του θέματος. Η χρήση νέων τεχνολογιών λοιπόν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, αυτό είναι κατανοητό, Από την άλλη, ναι, μεν παραβιάζεται περισσότερο το δικαίωμα της ιδιωτική ζωής από το τρέχον σύστημα που χρησιμοποιούμε η τεχνολογία αυτή τη στιγμή και ε, θεωρούμε όμως ότι υπάρχει περιθώριο για να γίνει μια κοινή απόφαση και να ληφθούν αποφάσεις συντονισμένα. Αυτά όλα πέραν των συζητήσεων που προκύπτουν γύρω από αυτή τη συζήτηση. Ε, κατά την άποψή μου, ορισμένα πράγματα που ακούμε είναι υπερβολικά. Όσον αφορά τώρα τις αεροπορικές υπηρεσίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις εργασίες της και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για το γύρο διαπραγματεύσεων που έχουν γίνει μέχρι τούδε. Έγινε ένας γύρος στη Washington, ένας ε, στη Μαδρίτη και εγώ θα βρίσκομαι και στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων που γίνεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές και η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι άνω του 60% της εναέριας κυκλοφορίας παγκοσμίω. Και αν υπάρξει άνοιγμα και τεχνικός και νομοθετικός συντονισμός θα δοθεί ένα σαφές μήνυμα στις υπόλοιπες ε, εναέριες αγορές. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα μειωθεί το κόστος, θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε καλύτερα την αλλαγή του κλίματος, διότι θα μειωθούν ε, οι χρόνοι των διαδρομών, ε, σημαίνει αυτό ότι μολύνουμε λιγότερο, ρηπαίνουμε ε, λιγότερο, γι' αυτό και με εκπλήσει και η άποψη του εκπροσώπου των Πρασίνων. Θεωρούμε ότι συνεισφέρουμε σημαντικά σε λιγότερες εκπομπές και στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Και υπάρχουν και πολλές πτυχές αυτής της συμφωνίας, ε, οι οποίες έχουν προχωρήσει. Έχουμε προχωρήσει πολύ τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον διότι εκεί ήδη υπάρχει μια κοινή θέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων και ελπίζουμε να προχωρήσουμε και στη δυνατότητα να επενδύουμε ε, αμφίδρομα και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το 25% το οποίο έχει καθοριστεί αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι υπάρχει καλή διάθεση από πλευράς Ηνωμένων πολιτιών, Έχουν δεχτεί να γίνει ένας τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και εγώ, χωρίς να είμαι υπερβολικά αισιόδοξο, θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο και για συμφωνία και για αλληλοκατανόηση. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε εντός δύο ημερών να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια νέα συμφωνία επί του θέματος αυτού. Όπως γνωρίζετε, η οδηγία για την ασφάλεια στους αερολιμένες ε, άρχισε να εξετάζεται το προηγούμενο εξάμεινο στο Συμβούλιο. Υπάρχει μεγάλη απόκληση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και επειδή ακριβώς ερίζουν οι απόψεις δεν έχουμε κατορθώσει μέχρι τώρα να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν καθορίζει πώς πρέπει να χρηματοδοτείται το θέμα της ασφάλειας στους αερολιμένες διότι κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό με διαφορετικό τρόπο σε εθνικό επίπεδο. Κάποιοι χρηματοδοτούν αυτά τα μέτρα μέσω ενός γενικότερου δασμού, ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι οι χρήστες ή οι επιβάτες αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ε, καταβάλουν τους φόρους για αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Για να καταλήξουμε λοιπόν σε συμφωνία στο θέμα αυτό, θα πρέπει ίσως να μην εστιάσουμε τη συζήτησή μας στην πηγή χρηματοδότησης για το φόρο, αλλά να εστιάσουμε σε αυτό που κατά την άποψή μου είναι ο βασικός αντικειμενικός στόχος αυτής της συζήτηση, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται, όπως είπε και κάποιος ε, συνάδελφος, μεγαλύτερη διαφάνεια και δεν θα επιτρέπει να γίνεται διάκριση στον καθορισμό αυτού του εφόρου στους ε, ρολημένες. Αυτός λοιπόν είναι ο προσανατολισμός που θα ε, προσπαθήσει να δώσει η Ισπανική Προεδρία. Μου μιλήσατε και για τις παρεξηγήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εγώ ε, πάντα έχω κανόνα μου ότι με το διάλογο καταφέρνουμε να κατανοήσουμε ένα τον άλλον και πιστεύω ότι μέσω διαλόγου θα κατανοεί και το ένα θεσμικό όργανο το άλλο. Τώρα, όσον αφορά στη χρηματοδότηση, ο στόχος ε, ο οποίος καθορίστηκε από την Ισπανική Προεδρία και το στόχο αυτό το συμμερίζεται και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι στη διάρκεια αυτή του χρονικού διαστήματος θα καθορίσουμε την ε, μεθοδολογία για την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Γι' αυτό ακριβώ και εργαζόμαστε πολύ εντατικά. Έχουμε ήδη συμμετάσχει σε ε, αρκετέ ομάδε εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να συζητήσει το θέμα τη αναθεώρηση. Δεν μπορώ να σα πω εκ των προτέρων ποια θα είναι τα κριτήρια για την αναθεώρηση, γιατί ακόμα εκρεμεί η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι να καθορίσουμε κάποια κριτήρια τα οποία θα τεθούν για τα διευρωπαϊκή ε, δίκτρια. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ε, και για τον καθορισμό των κριτηρίων, φιλόδοξοι και για την ε, διεύρυνση των διευρωπαϊκών μας δικτύων ε, η χώρα μου έχει και τη δική της φιλοδοξία σε αυτή την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων, την οποία συμμερίζεται και με άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να δοθεί μία ε, όθηση για αυτό τον ε, ε, διάδρομο της Μεσογείου, που δεν είναι ένας διάδρομος, θα είναι μία απόδειξη ότι μπορούμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών, το οποίο κατά την άποψή μας είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προωθούμε τη σήμερον ημέρα. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, δύσκολης οικονομικής κατάστασης, γι' αυτό και ακριβώς ε, ε, δυσκολεύουν και τα κριτήρια επενδύσεων. θα υπάρξει μια ημερίδα ε, ημέρες RTNT ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και εκεί θα καθορίσουμε και τη στρατηγική αναθεώρησης καθώς επίσης ε, πέραν από τη στρατηγική χρηματοδότηση θα συζητήσουμε και το βαθμό ε, προόδου των διαφόρων προγραμμάτων λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την εξωτερική διάσταση των διευρωπαϊκών δικτύων και τις σχέσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την ενσωμάτωση όλων των ε, υπηρεσιών μεταφορών. Η κυρία Μπιλμπάου μου έκανε μία ερώτηση η οποία ε, υπερβαίνει τα εσωτερικά θέματα της ε, χώρας μας και είναι μία ερώτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μία διακυβερνητική απόφαση των κυβερνήσεων δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει ένα διεθνές τμήμα σε κάποιο διάδρομο ε, στις επόμενες εβδομάδες, τον Απρίλιο, θα γίνει μια συνεδρίαση με τη Γαλλία για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε οριστικά για το διεθνές τμήμα του διαδρόμου. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεδρίαση και όταν θα συμφωνήσουμε και μεταξύ των δύο χωρών για το διεθνές αυτό τμήμα, θα μπορέσω να σας απαντήσω στην ερώτησή σας. Συνήθως δεν ε, προλαμβάνω καταστάσεις, απαντώ όταν υπάρχει κάτι οριστικό, κάτι σαφές και έχουμε καθορίσει τα κριτήρια. Με ρωτήσατε το θέμα ε, της Ευρωβινιέτας. Να πω ότι έχω απαντήσει στο θέμα αυτό και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ. Θα σας δώσω την ίδια απάντηση. Ναι, θα γίνει μια τεχνική συνεδρίαση στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας όπως ακριβώς δεσμεύτηκα όταν ήρθα εδώ στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Όσον αφορά τώρα στα δικαιώματα των επιβατών σε λεωφορεία και σιδηροδρόμους, να σας πω ότι η ανταγωνιστικότητα των μέσων μεταφοράς ε, πηγαίνει χέρι-χέρι με την ποιότητα των υπηρεσιών και αυτές πηγαίνουν χέρι-χέρι με την διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών. Γι' αυτό λοιπόν τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν θαλάσσιες μεταφορές, όπως επίσης και όσοι χρησιμοποιούν λεωφορεία ε, ή σιδηροδρόμους αποτελεί προτεραιότητα για την Ισπανική Προεδρία. Όπως σας είπα στις 11 Μαρτίου στο Συμβούλιο, υιοθετήθηκαν κάποιες θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για αυτές τις δύο σημαντικές προτάσεις, οι οποίες στόχο έχουν να ενισχύσουν τα δικαιώματα των επιβατών σε λεωφορεία, σιδηροδρόμους και σε πλοία, ε, και στη θάλασσα και στις ε, ποτάμιες οδούς. Ε, και θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με το Κοινοβούλιο, όπως ακριβώς υποχρεώμαθε, εντό σύντομου χρονικού διαστήματος, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό τον κανονισμό από κοινού για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Την επόμενη εβδομάδα πήγα να πω, όντως την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια συνεδρίαση μιας διάσκεψης υψηλού επίπεδου. Ελπίζω η παρουσία της Ισπανικής Προεδρίας να καταδείξει πόσο σημασία δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα θέματα. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει υψηλό επίπεδο συμμετοχής σε αυτή τη διάσκεψη και Για το θέμα αυτό η Ισπανική Προεδρία θα κάνει προσπάθειες προκειμένου να υπάρχει μία πιο αποφασιστική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της ασφάλειας, να λαμβάνεται υπόψη το θέμα της κατάρτισης των πιλότων, αναθεωρώντας και εξυγχρονίζοντας τις μεθόδους ε, στο πιλωτήριο, ε, αυξάνοντας την ανταλλαγή δεδομένων, δίνοντας μια κάποια όθηση για τις ε, διεθνείς σχέσεις ε, των ε, αεροπορικών εταιριών και των ασφαλιστικών εταιριών, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες στους επιβάτες και αναπτύσσονταν και κάποιες νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση μέσω δορυφόρου των αεροπλάνων βάσω του προγράμματος ΣΕΖΑΡ. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στο θέμα του ενιαίου ουρανού. Στην ε, συνεδρίαση της Μαδρίτης έγινε μια πολύ σημαντική δήλωση με πάρα πολλές ε, συστάσεις οι οποίες είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν στην, ε, κατά την έναρξη ισχύω του ενίου ουρανού και όλα αυτά περιλαμβάνονται στη δήλωση. Είμαι βέβαιος ότι όταν θα εφαρμοστεί αυτό το δεύτερο πακέτο στο νομοθετικό πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από ενιαίο νόμισμα και ενιαία αγορά, θα έχουμε και έναν ενιαίο ουρανό που θα μας δώσει τη δυνατότητα και σε εμά και στις ευρωπαϊκές μας εταιρείε να προσφέρουν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες, να έχουμε λιγότερες καθυστερήσεις για τους επιβάτες, να υπάρχει μια σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και μια σημαντική αύξηση της ασφάλειας. Η Προεδρία μελετά τη δυνατότητα, αυτό το έθεσε και η κυρία Χιάλα, να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών ε, τον Ιούνιο μία συζήτηση για τη στρατηγική για το 2020 υπό την προοπτική των μεταφορών και των επιπτώσεών τους ε, στην καινοτομία, στην απασχόληση και στην οικονομική ανάκαμψη. Κυρίες και κύριοι, σίγουρα κάποιες από τις ερωτήσεις που μου θέσατε δεν μπόρεσα να τις απαντήσω. Δυστυχώς ε, μας πιέζει ο χρόνος, έπρεπε να είχα ολοκληρώσει πριν από 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους ε, για όλα όσα άκουσα. Σημειώνω τις ερωτήσεις ε, που μου διατυπώθησαν και δεν μπόρεσα να απαντήσω και θα απαντήσω γραπτό στους βουλευτές στις, σε όλες τις ερωτήσεις που δεν πρόλαβα να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που για μία ακόμα φορά ξαναήρθατε να μας μιλήσετε όπως είχατε πει ε, ούτως ή άλλως στην αρχή της ε, θητείας σας ας πούμε, στην αρχή της Προεδρίας και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, Ισπανική Προεδρία γιατί βλέπουμε ότι γίνεται πολλή δουλειά και όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και όσον αφορά και άλλα θέματα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το διάλογο με εσά και την ομάδα, σας, την ομάδα σας όπως ας πούμε δικαιώματα των εργαζομένων ε, προστασία των εργαζομένων στην, ε, ε, στην αυτιλία, ασφάλεια μεταφορών, την μεταφορά φορτίων με το σιδηρόδρομο, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Επίσης, βασιζόμαστε και στην βοήθειά σας όσον αφορά τη στρατηγική 2020. Βεβαίως στη Σαραγώσα περιμένουμε ότι θα γίνει πολύ σοβαρή συζήτηση και δουλειά. Θα είμαι και εγώ εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. We just have minutes to... Πέντε λεπτάκια λέει ο Πρόεδρος έτσι ώστε να βάλουμε όλα αυτά τα ε, gadgets, τα τεχνολογικά τα οποία ε, χρειάζονται για την επόμενη παρουσίαση. Λίγη υπομονή λοιπόν. Okay, colleagues. Next item on the agenda is the 10 financing. Λοιπόν, το επόμενο σημείο της ημέρας έδεξης είναι η ανταλλαγή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σχετικά με τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Έχουμε τον κύριο Γιούκα Λούκαναν από την Φιλανδία που είναι τμήματάρχης της ε, διορθωτικής ε, χρηματοδότησης των ε, να είναι το μόνο φιλανδικό όνομα που ξέρω. Δεν ξέρω το δικό σας το είπα σωστά ή όχι. Κύριε Λούκανεν, λοιπόν, παρακαλώ. Thank you, Chairman. Chairman, um, members of the... Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά ε, που βρίσκομαι μεταξύ σας και μπορώ να σας μιλήσω για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη χρηματοδότησή τους. Να σας υπενθυμίσω λίγο τι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων. Είναι απλά η, Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι η τράπεζα η οποία είναι ε, είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι Υπουργοί Οικονομικών ε, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ το Διευθυντικό Συμβούλιο αποτελείται από κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπα και προηγουμένως, ο στόχος μας είναι βεβαίως οι προτεραιότητες και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους κεντρικού στόχους είναι ακριβώς τα διευρωπαϊκά δίκτυα που αποτελούν και το θέμα μας σήμερα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν όσον αφορά την υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Υπάρχουν πολλές ε, πράσινες γραμμές εδώ αλλά και κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Πρέπει να πω δηλαδή ότι πολλά έχουν γίνει, ε, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, πολλές επενδύσεις, αλλά και σημαντικές επενδύσεις εξακολουθούν ακόμα να πρέπει να ε, υλοποιηθούν. Οι ανάγκες ε, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στην περίοδο 2007-2013 η ανάγκη χρηματοδότησης είναι 390 περίπου δισεκατομμύρια. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση. Είναι πολλαπλές οι πηγές μια και πρόκειται για τόσο μεγάλα ποσά και επομένως, έστω και αν οι ε, πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φτάνουν να καλύψουν ένα περίπου 30% της απαραίτητης χρηματοδότησης, παραμένει μεγάλο ποσοστό που θα πρέπει να καλυφθεί από το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Όπως είπα και προηγουμένως, τα ποσά είναι πάρα πολλά. 15 ε, ε, με 20% ε, των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2005-2009. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσό. Να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Εάν δούμε τώρα ε, στη, αν δούμε τώρα την υλοποίηση, βλέπουμε ότι ε, ακολουθεί μια αυξητική τάση. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει επίσης και μια σταθερή αύξηση της δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά το, τα TENS. E. και πρέπει να πω ότι πέρα από τα TENS e και τα PPP είναι αυτά τα οποία απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό της δανειοδότησης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 ε, επίσης ε, βλέπουμε ότι μέσω, από, μέσω δομημένων ε, χρηματοδοτήσεων διευκόλυνσης έχουμε χρηματοδότηση δανείων καθώς επίσης και την εγγύηση δανειοδότησης όσον αφορά συγκεκριμένα προγράμματα. Βεβαίως μέσα στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων προσπαθούμε να προλάβουμε και κάποιους κινδύνους όσον αφορά τα προγράμματα TENS. Ε, επίσης γίνονται επενδύσεις σε equity ε, funds και επίσης χρηματοδοτήσεις μέσω του λεγόμενου ε, χρηματοδοτικού οργάνου Μαργαρίτας και φυσικά χρηματοδοτούμε σε μεγάλο μέρος και το ECTF. Τα τελευταία χρόνια ε, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί ιδιαίτερα σε αυτές τις συμπράξεις δημοσίου και ε, ιδιωτικού τομέα, αυτά τα ε, PPPs. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα, περίπου 120 προγράμματα PPPs και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη υπογραφές οι οποίες περνούν τα δύο δις. Όσον αφορά τώρα τις ολοκληρωμένες διαδικασίες PPP, εδώ σας έχω ένα κατάλογο ε, ε, ε, προγραμμάτων τα οποία στηρίξαμε το 2008 και το 2009 έτσι ώστε μπορείτε να δείτε εδώ και κάποια γνωστά ονόματα. Και βεβαίω το ποσό το οποίο βλέπετε στα δεξιά κάθε υλοποιημένου προγράμματος αφορά την δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα ήθελα πάρα πολύ ε, σύντομα να αναφερθώ σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή ε, την δομημένη διευκόλυνση χρηματοδότησης, το SFF. Ε, εδώ ε, κάνουμε δανειοδότηση και χρηματοδότηση ακόμα και κάτω από την αποδεκτή γραμμή ε, δανειοδότησης και πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τα SFF είχαμε 4,2 δισεκατομμύρια για το 2008 και 5,8 για το 2009. Υπάρχουν όμως και κάποια πιο εξεζητημένα προγράμματα όσον αφορά τα TENS. Το LGTT ας πούμε είναι ένα ιδιαίτερο ιδιαίτερα αποτελεσματικό ε, εργαλείο. Πρόκειται για ε, ε, ένα εργαλείο το οποίο δίνει την δυνατότητα επιπλέον ανάληψης κινδύνου και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο λαμβάνοντας υπόψη την ασάφεια των αγορών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως να βοηθήσουμε τον ε, ε, δημόσιο τομέα ε, να αντιμετωπίσει αυτές τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τα PPPs. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το European PPP Expertise Center, το οποίο βοηθάει έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες ε, ε, γνώσεις και να μεταφερθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία. Πάντα όσον αφορά την τεχνική αρρωγή έχουμε το JESPERS. Ο ρόλος του Jaspers λοιπόν βεβαίως που αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της Τράπεζας, ε, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακών ε, Θεμάτων, της BERD ε, και της KFW, είναι να διευκολύνει την χρήση και την απορρόφηση των πόρων των διαθετικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για το 2007 μέχρι το 2013. Το European Clean Transport Facility, ECTF, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την απόψή μας. Only lent ε, είχα πει προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, επίσης ε, κάνει επενδύσεις σε equity funds. Βλέπετε εδώ ένα κατάλογο που μας δείχνει την ευρεία γεωγραφική κατανομή αυτών των equity funds που ξεπερνούν το μισό δις που ενδεχομένως σα φαίνεται λίγο σε σχέση με τι ε, συνολικέ δυνατότητε χρηματοδότηση, αλλά που σα βεβαιώνω ότι είναι ένα πάρα πολύ, τη τράπεζα, αλλά σα βεβαιώνω είναι ένα πάρα πολύ ε, ψηλό ε, ποσό. Αναφέρθηκα προηγουμένω στην Μαργαρίτα. Είναι αυτό το ταμείο για την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την υποδομή για το 2020 το Margaret Fund, αυτό το ταμείο της Μαργαρίτας, ε, είναι ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό ταμείο, το οποίο χρηματοδοτείται από την τράπεζα, το CDC, το CDP, το ICO, το PKO και το KFW. Όμως, παραμένουν σημαντικές ανάγκες. Παρά τις πολλές προσπάθειες αλλά και τις πολλές επιτυχίες, δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε διαρκώς το μέλλον. Δύο μεγάλα θέματα ε, αναδύονται τα ε, προγράμματα είναι τόσο σημαντικά που η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα φαίνεται ε, επιβεβλημένη. Και η διευκόλυνση ιδιωτικής χρηματοδότησης των TENS φαίνεται να είναι απολύτως απαραίτητη. Βεβαίως ε, ο τομέας ε, των ε, μεταφορών θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιήσει τις γνωστές τεχνολογίες, καινούργιες τεχνολογίες έτσι ώστε να αναπτυχθεί αλλά ταυτόχρονα να είναι πιο φιλικός προς το χρήστη αλλά και πιο φιλικός προς το περιβάλλον, πιο πράσινη δηλαδή ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, είναι ε, να διευκολύνει και επιπλέον ε, επενδύσεις όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, να καθορίσει equity funds έτσι ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση της υποδομής των δικτύων όπως ας πούμε το Ταμείο της Μαργαρίτας για το 2020 να βελτιώσει τον συντονισμό των ταμείων και των πόρων που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ότι θα πρέπει να διευρυνθούν οι επενδύσεις μέσα από, μέσα από ε, θεσμούς ε, ε, κεφαλαιακούς και χρηματοπιστωτικούς. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η διευκόλυνση, η διευκόλυνση έκδοσης ομολόγων μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μηχανισμό. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να εφαρμόζεται η βαθμονόμηση αυτών των ομολόγων είναι σημαντικό να ε, χρησιμοποιηθεί σωστά το εργαλείο αυτό έτσι ώστε να έχει καλό αποτέλεσμα ε, και ένα μικρό ε, αρχικό ποσό μπορεί να επιτρέψει στις αγορές να χρηματοδοτήσουν μέσω ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης το εργαλείο αυτό και βεβαίως να υπάρξει ε, καταμερισμός του κινδύνου, έτσι ώστε να γίνει και πιο ελκυστικό σαν εργαλείο. Ένα άλλο σημαντικό ε, θέμα θα ήταν η διευκόλυνση ε, της έκδοσης ομολόγων μέσω παροχής εγγύησεων. Δηλαδή, αντί για δανειοδότηση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να παράσχει εγγύησεις με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λιγότεροι πόροι της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης και επομένως το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό με χρήση λιγότερων κονδυλίων από πλευράς του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου του εφαρμογής του LGTT, αυτό το εργαλείο, το LGTT, είναι ε, σχεδιασμένο ακριβώς έτσι ώστε ε, να ε, μπορεί να βρει ενδιαφερόμενους μέσα από ένα πολύ ευρύτερο φάσμα υποψηφίων. Και νομίζω ότι όλες οι πλευρές διεύρυνσης, οι δυνατότητες μάλλον διεύρυνσης του LGTT θα πρέπει να μελετηθούν. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα μπορούσαμε μέσω της διεύρυνσης του πεδίου του LGTT να ε, ε, ε, στοχοθετήσουμε πολύ πιο μεγάλες και περισσότερες επενδύσεις όσον αφορά τους υδροδρόμους αλλά και όσον αφορά τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τελευταίο αλλά όχι ελάσσον όπως συνηθίζεται να λέμε, είναι η δυνατότητα βελτίωσης ε, του συντονισμού των ε, πόρων και των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως ε, το, ε, ο προπολογισμό ε, των διευρωπαϊκών δικτύων και το Ταμείο συνοχή είναι ε, τα ταμεία τα οποία περισσότερο στηρίζουν από κοινωτική απόψεω την εφαρμογή των προγραμμάτων TENS. Και επομένω είναι σημαντικό να έχουμε διαθέσιμους πόρους και να είμαστε πάντα σε θέση να ανταποκριθούμε στι ανάγκε που παρουσιάζονται. Αυτά είχα να σα πω. Τώρα βλέπετε εδώ ένα πίνακα με τα τηλέφωνα και τα email των ανθρώπων με τους οποίους μπορείτε να έρθετε σε επαφή και βεβαίως μπορείτε να μου θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα. Thank you very much indeed, Mr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λούκανεν. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ειλικρινά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αλλά δεν κανένας εκ των έσω η παρουσίαση αυτή ήταν κάπως περίπλοκη. Από ό,τι κατάλαβα στα διαφορετικά δίκτυα προηγουμένω, τα πράσινα ήταν σωστά, τα κόκκινα ήταν, δεν ήταν καλά. Αυτό το κατάλαβα, μου φαίνεται, μέχρι εκεί. Αυτό που σας ενδιαφέρει εδώ, ιδιαίτερα, στο Κοινοβούλιο, και προσωπικά εμένα, είναι να ξέρω πώς μπορούμε αύριο να δημιουργήσουμε χρηματοδοτικά μέσα που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη ή θα τους δίνουν ισχυρότερα κίνητρα για να προωθήσουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα εφόσον καθοριστούν επιτέλους οι προτεραιότητες. Στο τέλος αναφερθήκατε σε κάποιες δυνατότητες της μεγαλύτερης παρέμβασης, αλλά κατά βάση, κατά τη γνώμη μου, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα. Σε μία σχέση 390 προς 270 και 270 είναι το υπόλοιπο, κατά πόσον για το μέλλον μπορούμε να έχουμε την ελπίδα ότι τα σχέδια αυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πιο γρήγορα και καλύτερα ή θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ισχυροί στην αρχή και τις να δώσουμε πιο ισχυρές γιατί στην πρώτη φάση ο κίνδυνος και για τον ιδιωτικό επενδυτή είναι πάρα πολύ μεγάλος Και γι' αυτό, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξέρω πώς προβλέπετε εσείς μια δυναμωμένη μορφή παρέγκασης με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν σήμερα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πολύ πιο γενικό. Κατά εδώ υπάρχει ένα σχέδιο από το Βέλγιο. Entrabel Rail Tunnel. Για το 2008 το έχετε το σχέδιο αυτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε συγκεκριμένα πώς εγγυηθήκατε την ιδιωτική συμμετοχή εκεί. Γιατί το έχετε στα PPP και PPP από όσο ξέρω είναι συμπραξή ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και θα ήθελα να ξέρω ο ιδιωτικός εταίρος εδώ πώς λειτουργήσε. Τελευταίο ερώτημα που έχω πάνω στην παρουσίασή σας. Είναι μια ερώτηση της οποια την απάντηση εν μέρη γνωρίζουμε. Πολλά χρηματοδοτικά μέσα έχασαν το δυναμικό τους λόγω της κρίσης φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όμως ε, είναι πιο ενδυναμωμένη με την κρίση σαν χρηματοπιστωτικός ε, φορέας στην αγορά. Πώς γίνεται αυτό, μήπως μπορείτε να δώσετε κάποιες ιδέες και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πώς θα μπορέσουν να σταθεροποιηθούν καλύτερα για να, μετά από αυτό που γνώσαμε στην Ευρώπη και στην Αμερική σε ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρός. Όπως βλέπετε κύριε Λουκάν, εκπροσωπείται πολύ καλά το Βέλγιο εδώ και μπορώ αμέσως να περάσω τον κύριο Αλκαντράουι, άλλος Βέλγος που θα μιλήσει τώρα και το ονόματος των σοσιαλιστών. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω αναφερθώ στην ε, ομιλία που ακούσαμε να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως. Να σας πω ότι ούτε και εγώ τα κατάλαβα όλα. Ε, πρέπει κάποιο να διαβάσει μάλλον αυτό το κείμενο μας, ώστε ε, εντάξει, κάποιες παρατηρήσεις έχω να κάνω όμως ήδη. Έχουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πρόκληση. Η δική μας επιτροπή, αλλά γενικά ο τομέας των μεταφορών και αυτό εν ώψη δυσκόλων χρηματοπιστωτικών καταστάσεων σε όλα τα κράτη-μέλη και πρέπει να γίνουν επενδύσεις που απαιτούνται και που μας κάνουν ε, να αναπτυχθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για μελλοντική ανάπτυξη. Αυτή η συζήτηση είναι τεράστια. Μπορούμε χρόνια να συζητάμε τι σκεφτόμαστε, ο Επίτροπος έχει κατά νου κάποιο ταμείο μεταφορών, αλλά εγώ σας ρωτάω εσάς, εσείς, τι θα συστήνατε. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό κατά τον δικότερο δυνατό τρόπο, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερους πόρους από εκείνοι που διαφαίνονται εκ πρώτης όψεως. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί εδώ που έχετε απαριθμίσει. αλλά αυτούς μπορούμε νομίζω αρκετά απλά να χρησιμοποιήσουμε. Και μία παρατηρήση ακόμα. Νομίζω το διάβολο είναι αυτό που αναφέρεται, αυτό που έφερε και ο κ αυτό που περνάει κάτω από το αεροδρόμιο των Βρυξελών. Οι ταξιδιώτες που θα περνάνε στο μέλλον κάτω από το αεροδρόμιο για να πάνε στο Λέβεν και στην Λιέχη θα πρέπει να πληρώνουν επιπλέον. Αυτό το θέμα βέβαια τίθεται. Και κάτι πιο συγκεκριμένο για τη Μαργαρίτα. Ε, Eh, Ποια είναι και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, πώς θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα σχέδια και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για το μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ότι και οι συνάδελφοι που είναι εδώ πιο πολύ χρονικό διάστημα στην Επιτροπή Μεταφορών δεν, κατάλαβαν τα πάντα γιατί και εγώ δεν κατάλαβα τα πάντα, χρειάζεται ίσως κανένας περισσότερο χρόνο. Συγκεκριμένα θέματα αναφέρατε διάφορα σχέδια που υποστηρίξατε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αντιβρίσεως στο PPP το 2008 και το 2009. Έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα σχέδια που μας παρουσιάσατε. Δεύτερον, ο Επίτροπος Κάλλας και στην ακρόασή του και όταν ήρθε εδώ μας είπε ότι Εκείνο θεωρεί τον τομέα των μεταφορών πάρα πολύ σημαντικό, φυσικό είναι αυτό, και για το μέλλον. Βέβαια, χωρί μεταφορέ δεν υπάρχει ε, ομαλή λειτουργία τη εσωτερική αγορά και θα πρέπει όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διάφορα κράτη-μέλη αλλά και στι περιφέρειε να δούμε ότι τα ταμεία ήταν άδεια και γι' αυτό δεν μπορούσαν καν να γίνουν οι τα απαραίτητα έργα συντήρηση των δρόμων και των συνδρομικών ε, εγκαταστάσεων. Γι' αυτό είπε ο κ. Καράς ότι θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε ε, μια νέα μορφή ταμείου εκτός από τα PPP. Φαντάζεσαι ότι υπάρχει ένα ε, μέλλον γι' αυτό. Γιατί όλοι οι διαφορά, όπως είπε και ο Σαρκαδρόη, τι θα μας πείτε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα χρήματα για τις μεταφορές. Τι μπορούμε να κάνουμε εσείς λέτε τι βοήθειες δίνετε, εμείς σκεφτόμαστε τι μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, όπως και άλλοι, την ίδια, την ίδια αντίδραση είχα. Ευτυχώς πέρσι τέσσερις-πέντε τραπεζίτες με εξήγησαν το θέμα της ε, χρηματοδότησης, ομολογώ ότι όλα αυτά δεν ε, μείωσαν τη φρίκη μου για όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί από ό,τι βλέπω αναβάλλονται τα χρέη προς το μέλλον και φτάνουμε σε ένα σημείο που τα κράτη δεν μπορούν πια να ε, αναποκριθούν στην εξυπηρέτηση του χρέους. Δυστυχώς έχουμε επίκαιρα παραδείγματα αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Μετά, όταν ο μηχανισμός ε, ε, επιλέγει τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και εσείς μας είπατε και για το 2008 και 2009 κάποια στοιχεία, τι γίνεται από το 2007 μέχρι το 2013 για όλη τη χρονική περίοδο. Γιατί αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, δηλαδή η χρηματοδότηση από την ε, ΕΤΕΠ ε, ε, ε, χρησιμοποιείται κυρίως από τις οδικές μεταφορές. Εμείς θέλαμε να ενισχυθεί περισσότερο ο συνδρομικός τομέας. Αυτό όμως αντιστρέφεται. Ακόμα και αν μέσα στα πλαίσια των δικτύων εμείς διαθέτουμε πολλά χρήματα για τη χρηματοδότηση του συνδρομικού τομέα, αλλά από την συγχρηματοδότηση της ΕΤΕΠ βλέπουμε ότι ωφελούνται κυρίω οι οδικές μεταφορές. Υπάρχει δηλαδή κάποια ανισορροπία δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Α, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω εγώ τουλάχιστον. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ει βάρο των συνδρομικών μεταφορών. Και αυτό σχετίζεται ακριβώ με το γεγονό ότι υπάρχουν αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία αφεντός προστατεύουν τον ιδιωτικό ε, επενδυτή από απώλειες, αλλά όχι το δημόσιο. Και αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει, γιατί για την μελλοντική δομή του τομέα των μεταφορών είναι αντιπαραγωγικό εάν ευνοούμε τον ένα τομέα και οι άλλοι τομείς υστερούν ακριβώς τώρα που έχει υπάρχει έλλειψη των πόρων στα δημόσια ταμεία, αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη. Έχετε κάποιες στρατηγικές που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε για να μην είναι τόσο έντονη αυτή η ανισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων του πεδίου των μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Γιάννησεν. Yes, uh, thank you. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ομιλητή. Η ερώτησή μου είναι απλή. Είπατε ότι θα χρειαστούμε περισσότερο ιδιωτικό κεφάλαιο. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό θα συμβεί αλλά θα ήθελα να ακούσω τι προσκόμματα βλέπετε εσείς ε, στις συμπράξεις σε δημοσιοδιωτικό τομέα στις υποδομές. Θεωρώ εξαιρετικό το να βλέπουμε ένα τέτοιο φάσμα μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν δεν δείτε και το τα όσα έχει κάνει η τράπεζα είναι εξαιρετική η δουλειά σας. Όλα καλά, αλλά το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Κατά με μπορεί να υπάρχουν και νομικά κολλήματα σε κάποιες ε, χώρες μέλη ή κάποια προβλήματα. Στη χώρα μου, στη Δανία, Το είδαμε όταν είχαμε την ε, ε, γέφυρα Freeman Belt. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι μεν για τους οποίους η Γερμανία δεν ήθελε να συμμετάσχει, αλλά ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να δεχτούν ε, το μοντέλο μιας δημόσιας επιχείρησης, μια επιχείρηση του δημοσίου, η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση και από εκεί και πέρα ο ιδιωτικός τομέας θα έπρεπε να καταβάλει τα υπόλοιπα για την γέφυρα. Ε, δεν είναι όμως θεωρίες, τελικά τα καταφέραμε, καταφέραμε να συνδέσουμε ε, με τη Σουηδία και κυρίως ο σύνδεσμος με τη Σουηδία ναι μεν ήταν δύσκολο στην αρχή αλλά αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Ε, Νομίζω ότι κάποια από τα νέα μέσα αναπτύχθηκαν ακριβώς από την Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύνδεση Σκανδιναβίας και Γερμανίας. Θεωρώ ότι τα ωφέλη ε, θα αφανούν στην πράξη. Θα ήθελα όμως να ακούσω κάποια ε, περισσότερα πράγματα για τα εμπόδια που υπάρχουν για τη συμπράξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ, κύριος Κράμερ μπορώ να σας πω δύο λόγια από τις δικές μου εμπειρίες. Για την γέφυρα αυτή στην Φέμαν Belt και την άλλη γέφυρα που είναι μεταξύ Κοπενχάης και μαλμό μεταξύ δύο μεγάλων πόλεων. Η άλλη όμως δεν εξυπηρετεί τόσο πολύ και θα πρέπει να, χρηματοδοθεί από τους χρήστες. Στην ε, Γερμανία πριν από 20 χρόνια όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσαμε την υποδομή μεταξύ ε, Ανατολής και Γερμανίας να την προωθήσουμε. Πολλά μπορούσαν, έπρεπε να γίνουν. Και τότε σκεφτήκαμε ότι χρειαζόμαστε αυτή την σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, γιατί αλλιώ δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτή είναι ομως μια κατάσταση που παρουσιάζεται μία φορά στον αιώνα, όπου είπαν ότι χρειαζόμαστε τώρα τεράστιες επενδύσεις για να μπορέσουμε να ενώσουμε τα δύο μέρη του, της χώρας. Ένα σχέδιο πραγματοποιήθηκε και μετά σταμάτησε. Γιατί, γιατί όταν εγώ σήμερα ε, δανείζομαι χρήματα που πρέπει να τα, ε, να τα επιστρέψω αργότερα, έχω αυτή τη στιγμή τεράστια κινητοποίηση πραγματο, παραδείγματος χάνει του τομέα ε, κατασκευών, το οποίο όμω ε, τελικά αποδεικνύεται ότι θα πρέπει να πληρώσω επί 10-20 χρόνια τα χρήματα αυτά χωρίς να έχω άλλα χρήματα για άλλες υποδομές. Δηλαδή έχουμε ε, μία έξαρση σύντομη και μετά τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από εκεί και πέρα. Μετά χρειαζόμαστε μία αλλαγή του τρόπου σκέπτεστε. Το είπα προηγουμένως ότι δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από τα μεγάλα προγράμματα που χρειάζονται 20 χρόνια να γεννήνουν και απορροφούν οι 80% των κεφαλαίων. Χρειαζόμαστε πιο μικρά σχέδια. Να έχουμε 80% ε, ας πούμε καλών υποδομών στην Ευρώπη και μετά να σκεφτούμε κάποιο μεγάλο σχέδιο. Τελευταία ερώτηση. Αυτά που είναι απαριθμισμένα εδώ. Βλέπω ότι το 90% είναι αυτοκινητόδρομοι. Μπορείτε να μου δώσετε αριθμητικά στοιχεία πόσο της 100 των χρημάτων χρησιμοποιούν οι εσωτικές μεταφορές, πόσο για τις συνδρομικέ ε, και πού αλλού τέλος πάντων θέλω να αναφερθώ στις μεταφορές με ποδήλατο, αλλά και εκεί υπάρχουν επιδοτήσεις. 50% των επενδύσεων θα πρέπει τουλάχιστον να χρηματοδοτούν τις συνδρομικές μεταφορέ αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουμε τους στόχους μας. Δηλαδή έχουμε μια πολιτική που διατυπώνουμε και οι οικονομικέ αποφάσεις κινούνται ακριβώς προ την αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί είδαμε τι έγινε στην Γερμανία και μια κυβέρνηση συντηρητική ε, τα κατήργησε όλα αυτά γιατί δεν υπήρχε καμία προοπτική. Ευχαριστώ κύριε Σπάλτσάκη. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų pateiktoje ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, πολλά αριθμητικά στοιχεία στην παρουσίασή σας και αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι οι υποχρεώσεις σας είναι 5 δις και αυτό που δαπανείτε εσείς είναι 500 εκατομμύρια. Και αυτό σχετίζεται και με τη μελλοντική πολιτική της τράπεζας. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν το εξή. Όταν πρόκειται να εξετάσουμε τις ε, προ... την ε, χρηματοδότηση των σχεδίων υποδομών, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στη χρηματοδότηση σχεδίων μεταφορών. Εσείς εδώ στο πίνακά σας έχετε πολλά σχέδια ενέργειας. Αλλά αν εμείς εδώ ασχολούμεθα με τις μεταφορές αγαθών και ταξιδιωτών, τότε θεωρώ ότι και η πολιτική μεταφορών και η πολιτική χρηματοδότηση των υποδομών θα πρέπει να επαναμελετηθούν για να μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Για τις πράξει ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα μου, είχαμε μια σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα για ένα σχέδιο στο Λονδίνο που ήταν η πιο σημαντική σύμπραξη που έγινε και ναι μένει στη θεωρία ακούγονται πάρα πολύ ωραία σε αυτές οι συμπράξεις αλλά η εμπειρία μου λέει ότι συνήθως το δημόσιο ε, έρχεται και κυριαρχεί, ενώ το ιδιωτικό κομμάτι είναι πιο περιορισμένο. Κάποιος έθεσε μια πολύ απλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν η κυρία Κένσεν ή η κυρία Μέσλερ. Έχω κι εγώ μια απλή ερώτηση να σας θέσω. Είναι πολύ ε, εύκολο να διατρέξουμε όλα αυτά τα σημεία τα οποία είχατε με τα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Εάν θέλω, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύσει χρήματα για το σιδηρόδρομο του Μάνσεστερ, Πώ θα τα καταφέρω. Και αυτό είναι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ στο κεφάλι μου το έχω πολύ καλά καθορισμένο και ξέρω πώς θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα και πώς ε, κάποια ε, μοντέλα μπορούν να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεις, κυρίως αν πρέπει να περάσουν ε, και από τις εθνικές κυβερνήσεις, το οποίο υποθέτω ότι πρέπει να γίνει. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι να συνεχίσω από αυτό που έλεγε ο Μάικολ. Εμένα με εξέπλεξε που είδα ε, πόσους αυτοκινητοδρόμους ε, και πόσες ότομπαν έχετε στο έγγραφο γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους. Αυτό νομίζω φαίνεται στα προγράμματα για το 2008-2009. Χαίρομαι που έχετε και κάποια τραμ και κάποιο μετρό, αλλά φαίνεται ότι οι περισσότεροι είναι αυτοκινητόδρομοι. Το οποίο νομίζω ότι ε, πηγαίνει αντίθετα στη θέση που ακολουθεί το Κοινοβούλιο σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για τη χρηματοδότηση των ΤΕΝ. Όταν λέτε ότι πρέπει να επενδύσουμε όλους μας τους πόρους, για παράδειγμα, στη χρηματοδότηση του ΤΕΝ. Εγώ μπορώ να το δεκτώ μεν αυτό, αλλά θα πρέπει να σέβεστε και τα ποσοστά τα οποία έχει καθορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τον καταμερισμό της χρηματοδότησης. Και αυτό με φέρνει στον ίδιο κύκλο. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε τον σιδηρόδρομο του Μάντσεστερ. να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πακέ από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο θα πει κάποια πράγματα από πλευρά του και μετά θα σα δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Κύριε Πακέ, παρακαλώ. Thank you. Thank you Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Δύο-τρία σχόλια. Να πω καταρχά ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται στενά και τα περισσότερα από τα μέσα αν όχι όλα τα μέσα που παρουσίασε ο κύριος Λουκάνεν σήμερα το απόγευμα, ήταν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επομένως, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη αλλά και τα εύσημα για αυτά τα μέτρα ε, και πολλά από αυτά σαφώς θα αναθεωρηθούν και ίσως και θα εξελιχθούν περαιτέρω, μπορεί και να αλλάξουν ε, στα πλαίσια της παρούσας συζήτησης ε, στην πολιτική αναθεώρησης του 10-10 Υπάρχει σαφώς η ανάγκη, το έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακρόασή της, το είπε και ο ε, κύριος ε, Λούτα σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική χρηματοδότησης για την εφαρμογή του δικτύου TEN10 και θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο και να έχουμε ένα πλαίσιο αποτελεσματικής επιλογής ε, στρατηγικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το θέμα φυσικά και της ισορροπίας θα ληφθεί υπόψη και θέλουμε να δούμε και τα διάφορα κονδύλια τα οποία διατίθενται για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ χρηματοδότησης και κονδυλίων και χρήστη και φορολογούμενου από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι οι δύο όροι μιας εξίσωσης όταν ε, βλέπετε τι γίνεται με τη στρατηγική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θα είναι κυρίως από πιστώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και από εκεί και πέρα οι επιπλέον επιδοτήσεις θα είναι ευθύνη των κρατών μελών και από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο βάρος μένει στα κράτη-μέλη. Η στρατηγική λοιπόν θα πρέπει να λάβει και αυτό υπόψη και να ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα πιο ε, στεναρό μοντέλο συντονισμού μεταξύ εθνικών επενδύσεων και ευρωπαϊκών επενδύσεων και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ε, μεταφορών και ίσως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μεταφορών να μπορούσε να εξυπηρετήσει και αυτό το, ε, το κομμάτι. Δεν μπορώ να σας εξασφαλίσω ότι τους επόμενους μήνες ε, θα προκύψει τόσο σαφώς αυτό, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει περιθώριο για περισσότερες επενδύσεις και υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης βέβαια. Πολλές ερωτήσεις που έθεσαν τα κράτη-μέλη είναι κυρίως πώς μπορούμε να έχουμε ε, πιο αποτελεσματικές υποδομές TEN 10. Ε, μπορείτε σίγουρα να κάνετε και εσείς συστάσεις και εμείς στην αναθεώρηση της πολιτικής μας θα εξετάσουμε όλους αυτούς τους τρόπους και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να δούμε δούμε πώς, κύριε Πρόεδρε, μπορεί όντως ο σιδηροδρόμος του Μάντσεστερ να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, διότι μπορεί να δοθούν δάνεια ή επιδοτήσεις μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών και να έχετε πολύ καλά προγράμματα στο δίκτυο του TEN10, τα οποία να μην... Ε, διατίθενται για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δηλαδή οι μηχανισμοί διασφάλισης, ε, όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και να δούμε και τι γίνεται με τις πράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι χρυσός κανόνας η σύμπραξη αυτή, τα PPP, όλοι το ξέρετε για τα TNT, τα... οι συμπράξεις αυτές είναι αποτελεσματικές γιατί ίσως σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι καλές, ε, μπορεί να έχουν πιο αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων και πιο αποτελεσματική διαχείριση. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν και επιπλέον χρηματοδότηση και επιπλέον έσοδα, αλλά οι συμπράξεις αυτές είναι περίπλοκες και σε περισσότερες, στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν στις δυνατότητες που έχουν θεσμικά τα κράτη-μέλη, οι τοπικές αρχές και πολλά πράγματα τα οποία ε, προφανώς είναι εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδατε και κάποια πράγματα στην ε, παρουσίαση του Γιούκα. Κοιτάμε να δούμε τι γίνεται με θεσμική ανάπτυξη και θεσμικές δυνατότητες, διότι είναι περίπλοκα τα θέματα αυτά και το θέμα στο τέλος τέλος είναι ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Και αυτό είναι ένα πολύ πολιτικό, πολύ περίπλοκο ζήτημα. Όλες οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι δύσκολα θέματα και γι' αυτό ακριβώς και δεν έχετε και τόσες πολλές όσο θα θέλατε να έχετε τελικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πακέ. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν. Ποιος αναλάβει τον κίνδυνο και νομίζω ότι... ο ιδιωτικός τομέας ε, τις περισσότερες φορές δεν θέλει να αναλάβει τον κίνδυνο. Τέλος πάντων, κύριε Λούκανεν, ε, έχετε μια-δύο ερωτήσει να απαντήσετε, θέλετε να απαντήσετε. Και αν, ε, αν θέλετε να δεχτείτε τώρα το σιδηρόδρομο του Μάντσεστερ, εγώ ευχαρίστως να σας ακούσω να το δέχεστε. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση να δω το, το θέμα του σιδηροδρόμου του Μάντσεστερ. Αρκετά ζητήματα εφήγησαν εδώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να τα καλύψω εν λεπτομερία όλα τα ζητήματα αυτά, γιατί είναι και περίπλοκα άλλωστε. Θα απαντήσω σε ορισμένα θέματα. Ένα θέμα το οποίο φαίνεται να επανέρχεται διαρκώς αφορά το γεγονός ότι δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση. Πώς λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με εξυπνότερο τρόπο τα χρήματα που έχουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε αντισταθμίσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εάν κανείς δει κυρίως ε, τις διαφάνειες που έδειξα προς το τέλος της παρουσίασής μου, ε, καταλαβαίνει ότι ε, το σημαντικό είναι να βρεθούν οι υποδομές αυτές οι οποίες θα διευκολύνουν την χρηματοδότηση των επενδύσεων και επομένως να γίνει όσο γίνεται περισσότερη δουλειά για κάθε επενδυόμενο ευρώ. Funding from EIB. Άλλα θέματα τώρα τα οποία θίξατε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οποιοδήποτε δανειστής μπορεί να απευθυνθεί βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και φυσικά από τη σειρά της η τράπεζα κάνει μια προεπιλογή μέσω μιας ε, διαδικασίας επιλεξιμότητας Το ίδιο γίνεται και έχει γίνει ήδη δηλαδή στην πρώτη φάση των TENS ε, ε, και βεβαίως μελετάται και η οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική ε, αηφορία, συγγνώμη, βιωσιμότητα του προγράμματος. Και φυσικά γίνεται και μελέτη όσον αφορά την δυνατότητα απόδοσης τη επένδυση, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρατε πολύ από εσά σχετικά με τα ε, προγράμματα 2008 και 2009 τα οποία ε, εμφάνισα ήταν κυρίως PPP ε, προγράμματα. Δηλαδή, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των, ε, ε, για τις μεταφορές. Δεν αφορούσε εξαντλητική παρουσίαση όλων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. και ε, τα χρήματα τα οποία ανέφερα αναφέρονται κυρίως στον τεχνικό διαχωρισμό. Στην τελευταία γραμμή της 7ης διαφάνειας δίνεται το ποσοστό της 100 των, ε, του συνόλου των ε, ε, διευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον σιδηρόδρομο. Βεβαίως υπάρχουν διακυμάνσεις τα διάφορα χρόνια. Και βεβαίως και στην χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων μπορούν να υπάρξουν διακυμάνσεις πρέπει να σας πω ότι στηρίζουμε κάθε μορφή μεταφοράς, αλλά κυρίως θέλουμε να προωθήσουμε αυτές τις μορφές που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Τώρα, αν με ρωτάτε αν λαμβάνουμε όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας στον προγραμματισμό που κάνουμε για το μέλλον, μπορώ να σας απαντήσω ως εξής. Ερώτηση εκτός μικροφώνου, δεν ακούν οι διερμηνείς δυστυχώς. Έχετε ένα ποσοστό ε, ε, ε, ένα ποσοστό της 100 για το ποια είναι τα, οι τρόποι μεταφοράς φιλική προς το περιβάλλον και ποιοι δεν είναι. δεν νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω πολύ διαφοροποιημένα στοιχεία. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσα να σας πω κάτι για τους σιδηροδρόμους, αλλά δεν αναφέρονται όλα εδώ. Ε, ε, υπάρχουν και οι θαλάσσιες μεταφορές κτλ. Όπως είπα και προηγουμένως, κάθε σχέδιο, κάθε πρόγραμμα το οποίο πρέπει να χρηματοδοτηθεί ή ζητά χρηματοδότηση, θα πρέπει να περάσει την προεπιλογή η οποία αφορά ακριβώς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Σχετικά με το μέλλον τώρα. Ένα ζήτημα το οποίο έθιξα είναι το, η, ενδεχόμενη διεύρυνση του στόχου του LGTT. Δηλαδή, είναι αυτό το κομμάτι που αφορά τις πιο πράσινες μεταφορές. Πρέπει να πω ότι δεν είναι πολλά τα προγράμματα συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου για το σιδηρόδρομο που να αφορούν τη διαχείριση κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να δούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρούμε τρόπους έτσι ώστε ε, να ανταποκριθούμε στις ε, υφιστάμενες ανάγκες έτσι ώστε να μπορέσουμε ας πούμε, να μπούμε περισσότερο σε κλάδους όπως είναι ο σιδηρόδρομος σχετικά με το Ταμείο της Μαργαρίτας. Πρέπει να σας πω ότι η Μαργαρίτα είναι ένα ανεξάρτητο ταμείο. με ανεξάρτητη συμβουλευτική, διαχειριστική και διοικητική δομή και επομένως οποιοδήποτε ενδιαφέρεται σε χρηματοδότηση από τη Μαργαρίτα σε, αυτά, σε αυτούς τους κεντρικούς ε, τομείς μπορεί να έρθει σε επαφή με τη συμβουλευτική ε, ομάδα και να ρωτήσει εάν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχουν τεθεί. Υπήρξε και μία ερώτηση σχετικά ε, με το κατά πόσον ο κατάλογος των PPPs που σας ε, υπέβαλα είναι εξαντλητικός. Όχι. Ε, στο κατάλογό μου αναφέρω άλλωστε μονάχα τα στοιχεία για το 2008 και 2009. Μία ερώτηση από την ε, ε, Δανέζα βουλευτή σχετικά με τα PPPs. Να σας πω το εξής. Ρεαλιστικός καταμερισμός κινδύνου. Μπορεί να είναι κοινότοπο, αλλά συνήθως λέμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αναλαμβάνεται από, το, από τον εταίρο αυτόν ο οποίος είναι καλύτερα σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διαχείριση κινδύνου. Ε, όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει μάλλον είναι συνηθισμένος να αναλαμβάνει κινδύνους, μόνο που ε, οποτεδήποτε αναλάβει περισσότερο κίνδυνο, χρειάζεται οικονομική διασφάλιση. Όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη η οικονομική διασφάλιση. Και βεβαίως, οποιαδήποτε ε, θετική εξέλιξη στο μέλλον θα μειώσει και το κόστος ε, διαχείρισης των προγραμμάτων. Και βεβαίως το σημαντικό είναι να καταλήξουμε τελικά σε κάποιες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες ε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιους οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ε, υπάρχουν επίσης χώρες οι οποίες κάνουν ε, μία σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και μετά τίποτα άλλο. Πρέπει να πω βέβαια ότι τα πρώτα πιλωτικά προγράμματα συνήθως είναι αυτά που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες και που είναι τα πιο δαπανηρά. Όταν όμως ε, οριστούν οι κάποιες ε, βέλτιστες πρακτικές, ε, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεπεράσει κανείς τις δυσκολίες. Και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση είναι και περισσότεροι οι ενδιαφερόμενοι από τον διεθνή χώρο. Και μπορώ να σας πω ότι για μελλοντικά σχέδια έχουμε αρκετούς ε, ε, ε, ενδιαφερόμενους που έχουν δηλαδή δείξει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για προγράμματα. Θα είδατε επίσης ότι συμπεριλαμβάνονται και ενεργειακά προγράμματα, το, το έγραφα στην διαφάνεια. Και βεβαίως η ενέργεια είναι μία από τις έξι προτεραιότητες που έχουμε. και βλέπετε ότι τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται όσον αφορά τις υποδομές περιλαμβάνουν και την ενέργεια δεν, και άλλα θέματα, δεν, είναι, δεν αφορούν αποκλειστικά τις ε, μεταφορές. Επίσης να σας πω ότι έχουν γίνει πολλές μελέτες σχετικά με τα μοντέλα ε, των ε, συμπράξεων ε, και το Γραφείο Οικονομικών ε, ελέγχων του Ηνωμένου Βασιλείου ε, έχει ε, διεξάγει τέτοιου είδους μελέτες. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. απλά το ανέφερα. Ανέφερα το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, νομίζω ότι απήντησα στι περισσότερε από τις ερωτήσει σα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Well, I don't want to open up a second or third or fourth. Δεν θέλω να ξεκινήσω δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο γύρο ερωτήσεων. Μπορείτε να κετέβετε όσο θέλετε. Είστε πολύ ωραία όταν κετέβετε. Θα σας επιτρέψω να παρέμβετε πολύ σύντομα για ένα σύντομο σχόλιο, αλλά αυτό ήταν. Κυρία Λίχτεμπεργκ. Αποφασίσαμε ένα κείμενο για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και εκεί αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα δίνει ξεκάθαρε τι πληροφορίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που πήραμε μέχρι στιγμή, ακόμα και η μία ακριβή απάντηση για την ερώτηση του 2010-2013, δεν είναι σύμφωνη με αυτό που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συνεργαστούμε σε άλλο επίπεδο. Γιατί ε, έχω βαρεθεί πια να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες λόγω της ε, χρηματοδοτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως δεν υλοποιούνται. Ευχαριστώ. Ο Μάικελ ένα λεπτό. Ναι. Είχα ρωτήσει τι θα γινόταν εάν τώρα τα επόμενα δέκα χρόνια πραγματοποιήσουμε πολλά προγράμματα και τα επόμενα χρόνια μετά πρέπει να τα επιστρέψουμε τα χρήματα. Γιατί θα παράγουμε ανεργία. Μια φυσαλίδα. Δεν απαντήσετε σε αυτό. Και αυτό το κριτήριο γιατί στη Γερμανία μια συνεργική κυβέρνηση σταμάτησε τις κοινοπραξίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Πρόεδρος, ωραία. Θέλετε να απαντήσετε? Όχι. I, I think I, I, um, Νομίζω ότι έκανα κάποιες παρατηρήσεις επί του θέματος. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Πακέ. ότι οι συμπράξεις αυτές δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση για όλα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει κάποιο όφελος για τα λεφτά που θα πανούμε. Εάν λοιπόν ε, μια τέτοια σύμπυραξη δεν είναι κατάλληλη για ε, μια συγκεκριμένη κατάσταση, τότε δεν είναι η μέθοδος μειοδοτικού διαγωνισμού που θα πρέπει να επιλέγετε. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι μιλήσαμε πάρα πολύ για τα PPP σήμερα, διότι είναι ένα από τα αναδυόμενα στοιχεία τα οποία έχουμε στην αγορά εν γέννη, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει όλες τις μεθόδους διαγωνισμών. Δεν έχουμε κάποια προτίμηση για τη μία ή την άλλη μέθοδο. τα παραδοσιακά ε, προγράμματα τα οποία προκύπτουν μέσω διαγωνισμών είναι αυτά στα οποία έχουμε τις ε, περισσότερες επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λούκανεν. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ε, μία εικόνα του τι κάνει ο Όσκαρ Λάινεν κάθε φορά στην πρώτη κατηγορία που προσπαθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις ε, των μελών. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις που δώσατε στα μέλη μας ε, και ακούσατε και τα όλα όσα είχαμε να σας πούμε. Ε, είμαι βέβαιος ότι η εικόνα που αποκομίσατε είναι ότι όλοι δεν πιστεύουν ότι είναι παράδεισος ε, οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι να υπάρχει πρόσβαση σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για πολύ σημαντικά προγράμματα μεταφορών και θέλουμε να τονίσουμε σε εσά ότι χρειαζόμαστε τέτοια πρόσβαση ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ιδέες μας ε, για όλα όσα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα για τις μεταφορές στην Ευρώπη και φυσικά αλληλένδετα με αυτά είναι και οι περιβαλλοντικές μας υποχρεώσεις και μειώσεις ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας ε, καλέσουμε εκ νέου κάποια στιγμή στο μέλλον και να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία συνάδελφοι. Να περάσουμε τώρα στα διάφορα. Δεν μου έχει πει κανεί κάποιος ότι έχει κάτι από τα διάφορα, εκτός αν θέλετε να θίξετε κάτι τώρα να σας πω ότι οι ημερομηνίε για την επόμενη συνεδρίαση είναι Δευτέρα 27 Απριλίου, 3 ε, η ώρα. Ελπίζω να σας ξαναδώ τότε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και την παθαρχία σας σήμερα το απόγευμα. Ε, τηρήσατε όλοι τα χρονικά περιφέρεια. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς ο Πρόεδρος και το προσωπικό για την επιτυχή διεξαγωγή της συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.